να προχωρήσουμε στη συνεδρίασή μας. Δεν είναι πολύ σωστό να προσκαλούμε κόσμο και να μην έρχεται κανείς από τους βουλευτές. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για τους ε, και καλεσμένους. Ίσως πρέπει να καλούμε λιγότερους ανθρώπους, αλλά να είμαστε παρόντες όταν έρχονται. Λοιπόν, δεν είναι τόσο ευχαριστά τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι έπρεπε να το πω τώρα. Έχω τη χαρά να χαιρετήσω τον κύριο Μαντελίν, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής τη ΣΥΝΣΟ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας και θα θέλαμε να ακούσουμε από σας και τους συναδέλφους για το σχεδιασμό στην Κομισιόν. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Κύριε Μαντιλένα, έχετε τον λόγο. Όχι, όχι. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, οφείλω να ομολογήσω ότι για μένα δεν μετράει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν ε, οι, οι προτάσεις ε, της Επιτροπής και του Επιτρόπου για τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές, και αυτό είναι καλό για όλους. Και ναι μεν καλό είναι να σκεφτόμαστε τι διακοπέ ε, αυτή την περίοδο, αλλά καλό είναι να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά τι διακοπέ. Εγώ θα κάνω κάποιε ε, παρατηρήσει ε, ε, παρατηρήσεις ε, και μετά ο συνάδελφό μου για, θα μιλήσει για το roaming, γιατί είναι καλό να ξέρουμε τι, είναι οι προτάσει μα για το roaming. Ας ξεκινήσουμε με τα θέματα της, διακυβέρνησης, της διακυβέρνησης και μετά πάμε στην, θα για την οικονομία. Η G8 στην Οντοβίλ πολύ καλά έκανε και, έκαναν και έθεσαν ε, τα θέματα του ίντερνετ στα, ε, σαν προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική καινοτομία, όχι για αυτό που αποφασίστηκε, αλλά γιατί το ίντερνετ και η διακυβέρνησή του είναι ένα πραγματικά κρίσιμο σημείο για όλο το οικοσύστημα του ίντερνετ. Και υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα ήθελα να θίξω εδώ και ξέρω ότι εσείς είσαστε εξοικειωμένοι. Κατα, καταρχάς το φόρουμ διακυβέρνησης του ίντερνετ που θα, ε, θα συναντηθεί για πρώτη φορά ε, μετά τη νέα θητεία στο Ναϊρόμπι το φθινόπωρο και ε, ευχαριστούμε γιατί τα μέλη του Κοινοβουλίου έκαναν κάποιες άτυπες συναντήσεις ε, για να προετοιμαστούν, να προετοιμαστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνει και πέρυσι στο Βίλνιους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχει, μια, υπάρχει ένα ενδιαφέρον πολυμερές, αν θέλετε, και όλοι θέλουμε να προχωρήσει το ίντερνετ. Δεύτερον, ίσως αυτό να μην είναι τόσο θετικό, βέβαια κατά την άποψή μου, είναι ότι ξεκινήσαμε στη συζήτηση με ε, ε, τους μεγάλους μας εταίρους για το ICAM. Όπως ξέρετε, από την τελευταία συνάντηση στο, στη Σιγκαπούρη. Το, ε, η ICAM έχει επιβεβαιώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην, για μια επόμενη θητεία. Ξέρετε επίσης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ανάλυσαν κάπως κάποια θέματα ε, σύγκρουσης των συμφερόντων γιατί το ICAM είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν και θετικά στοιχεία και λιγότερο θετικά, γιατί το ίντερνετ είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέα για όλους μας. Δεύτερον, όσον αφορά την ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας ε, προχωρήσαμε σημαντικά με τα κράτη-μέλη και στην άτυπη Υπουργική Συμβου... στο ε, Συμβούλιο στον Πάλατον, αλλά και στην, ε, στο... στην Υπουργική Σύνοδο για να ε, αυξήσουμε την ασφάλεια όλων των χρηστών του ίντερνετ, πολιτών, εταιρείων, επιχειρήσεων, ε, ε, εκπροσώπων των δημόσιων υπηρεσιών και βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές επιθέσεις και από hackers σε, στο Υπουργείο Εμπορίου της Γαλλίας, στην, σε δημόσιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, η απειλή αυξάνει όσον αφορά την ασφάλεια, όπως είχαμε για το SARS και για την ε, γρήπη των πουλερικών. Ε, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει, καταρχάς να δημιουργηθεί ένα όραμα πιο ενεργών ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, δηλαδή να υπάρχει μια συλλογική δράση από πλευρά των κρατών μελών και κατά δεύτερον υπάρχει και μια πρόταση στον προϋπολογισμό για την ε, σύνδεση, αν θέλετε, του, της Ευρώπης. Συνήθως όταν μιλάμε για σύνδεση εννοούμε για την ευρεία ζώνη, για, τους, ε, για τις λεωφόρους, ε, τις τεχνολογίες ή τις λεωφόρους γενικότερα, τους αυτοκινητοδρόμους, αλλά εμείς μιλάμε για συγκεκριμένη σύνδεση, για καλώδια, για τα υδραυλικά τέλος πάντων, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Και στην ΙΖΑ όχι μόνο ανανεώνουμε την θητεία, αλλά ε, συνεδριάζουμε και με το Συμβούλιο για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, έθιξα το θέμα της έρευνας, όπως είπαμε και προηγουμένως, λέγαμε προηγουμένως πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, είναι δύσκολη καιρή για την δημόσια χρηματοδότηση. Και η Κομισιόν πιστεύει ότι η πρόταση για μια σημαντική αύξηση όσον αφορά τις δαπάνες στην έρευνα και στην ανάπτυξη και την καινοτομία χρειάζεται, αν θέλετε συν 46% από το FP7 και στις προτάσεις που είχαμε. Δεν είναι πολυτέλεια η αύξηση αυτή. Ε, πιστεύω ότι και εσείς και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούμε. Από τη δική μου σκοπιά, τη μικρή σκοπιά αν θέλετε της έρευνας, πιστεύουμε ότι η μεσοπρόθεσμη εκτίμηση αυτών των οποίων κάνουμε, πιστεύουμε ότι κάθε ευρώ του φορολογούμενου το δαπανούμε με τον σωστό τρόπο. Και θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να το, να το καταλαβαίνουν και οι συνάδελφοί σας ότι όντως ξοδεύουμε σωστά τα ευρώ. Προτείνουμε στο μέλλον οι, προ, οι προσπάθειες για την έρευνα είναι και μεγαλύτερες αλλά και μικρότερες. Δηλαδή θέλουμε τις ε, μικρές αν θέλετε τις γρήγορες ε, ε, προτάσεις που λειτουργούν γρήγορα και που αποδίδουν γρήγορα ε, έχουμε μικρές ιδέες ε, που μπορεί όμως ε, να είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά και οι μεγάλες αν θέλετε ιδέες και αυτές είναι χρήσιμες και αναγκαίες. Είδαμε ότι στον τομέα του ICT μπορούμε να, να έχουμε μια χρηματοδότηση, ένα κονδύλι ενό εκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια, εάν και, εντοπίσουμε, αν και εφόσον εντοπίσουμε δηλαδή σημαντικές δραστηριότητες που μπορούν να μας ε, εξασφαλίσουν μία πρόοδο. Επίσης είπαμε τη σύνδεση της Ευρώπης που είναι νέα πρόταση στον προπολογισμό, δεν ανήκει μεν στον τομέα της έρευνας αλλά πιστεύω ότι εμπίπτει στον ε, τομέα των δραστηριοτήτων ε, αυτής της Επιτροπής. Υπάρχει το, το πρόγραμμα ΖΕΟΝ, e είναι δηλαδή το δίκτυο το οποίο επιτρέπει στους Ευρωπαίου επιστήμονε επιστήμονες ε, να δουλεύουν με στην Ευρώπη με στοιχεία που δίνει το μεγάλο τηλεσκόπιο από την Χιλή ας πούμε και μετά όσον αφορά την οικονομία για τις τηλεπικοινωνίες που είναι και το κομμάτι που με αφορά όσον αφορά την οικονομία το πακέτο για την μεταφορά προχωράει πάρα πολύ σιγά ε, όλοι θα πρέπει να μεταφέρουν την νομοθεσία ε, άμεσα και πρέπει να ανησυχούμε, Πρόεδρε, γιατί ε, δεν έχει γίνει μετάθεση της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη και, και θα έλεγα ότι είναι πολλά τα κράτη-μέλη που δεν έχει γίνει αυτή η, μετα, η μεταφορά. Τώρα, μιλάμε για τις συστάσεις και όχι για την νομοθεσία αυτή καθεαυτή. Αν, αν δείτε τις συστάσεις ε, υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο θα ε, δημοσιευθεί το επόμενο διήμερο και που λέει ότι το ποσοστό της νομοθεσίας στην Ευρώπη ε, που στηρίζεται αν θέλετε στις συστάσεις μας πρέπει να βελτιωθεί. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει μια ευθυγράμμιση στον τομέα των επενδύσεων και στα κριτήρια για τις επενδύσεις. Άρα για τις ε, τηλεπικοινωνίες και την νομοθεσία για τις των τηλεπικοινωνιών πρέπει να γίνει ε, μια πρόοδος. Τώρα, για την πρόταση όσον αφορά το Ρόμι, και εδώ θα δώσω το λόγο στον αδελφό μου, η πρόταση για το Ρόμι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ε, γιατί ακριβώς εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του τοπίου για την ε, νομοθεσία της, των τηλεπικοινωνιών σαν ένα σημείο κορυφής αν θέλετε, σαν ένα πολύ σημαντικό σημείο, σαν την αποκορύφωση της νομοθεσίας. Και η πρόταση την οποία υποβάλλουμε είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά την, ε, τις διαδροτικές ε, αλλαγές και όχι απλώς και μόνο έναν έλεγχο των τιμών. Ε, παρακολουθούμε τις τιμές βέβαια και ε, από την ομιλία και το, MSS, και το SMS συγγνώμη, θέλουμε να καλύψουμε και τα δεδομένα. Άρα πρόκειται για ένα κομμάτι της νομοθεσίας το οποίο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Και εγώ στις διαφάνειες θέλω να, με τις διαφάνειες που θα σας δείξω, έχω σε στόχο να σας εξηγήσω τι ακριβώς προτείνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής. Προτού όμως φτάσω στο σημείο αυτό θέλω να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα ποια είναι η τωρινή κατάσταση και ποια είναι η μορφή της αγοράς σήμερα. Όπως αναφέρει λοιπόν ο τρέχον κανονισμός για την περιαγωγή, η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να, να αναθεωρήσει από τη βάση των εξελίξεων τον κανονισμό αυτό και σαν τμήμα αυτής της ε, αναθεώρησης και επισκόπησης καταλήξαμε σε μια έκθεση ως Κομισιόν η οποία περιλαμβάνει την προηγούμενη εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει μια δέσμη προτάσεων για τον κανονισμό της περιαγωγής του roaming δηλαδή στη συνέχεια. Αν δείτε τώρα την αγορά και τη μορφή που έχει πάρει και τον αντίκτυπο της τρέχουσας ρύθμισης του τρέχοντος κανονισμού. Είδαμε ότι γενικά υπήρξε ικανοποιητική συμμόρφωση των ε, παρόχων υπηρεσιών με τα τιμήματα για την περιαγωγή έχουν μειωθεί φυσικά και οι τιμές έχουν μειωθεί αλλά είναι πολύ κοντά στα άνω όρια. Αν δούμε την περιαγωγή δεδομένων, είναι μια αγορά η οποία αυξάνεται, είναι η ίδια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αγοράς του roaming, αλλά περιμένουμε να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Στον τρέχοντα κανονισμό, εμείς έχουμε ρυθμίσει την αγορά χονδρικής για τα δεδομένα και εδώ βλέπουμε να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός είναι 50 cent το, η οροφή για την περιαγωγή δεδομένων σε χοντρικό επίπεδο, αλλά αν δούμε τις τιμές λιανικής, ξεπερνούν κατά πολύ την τιμή χονδρικής. Αυτό το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει αυξηθεί το περιθώριο μεταξύ χονδρικής και λιανικής, δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών βγάζουν πολλά λεφτά από την παροχή υπηρεσιών. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια συγκεκριμένη μορφή συσχετισμού μεταξύ κόστους και τιμήματων. Έχω να σας δείξω δύο διαφάνειες εδώ για την τιμή περιαγωγής φωνητικής τηλεφωνίας, το κόστος του roaming και εδώ βλέπετε με σαφή τρόπο ότι υπάρχει πραγματικά ένα χάσμα και οι στήλες που βρίσκονται στο ύψος της διακεκομένης γραμμής δείχνουν το τι ακριβώς κυκλοφορεί στην αγορά σήμερα σαν τιμές ε, περιαγωγής. Και είναι πολύ κοντά λοιπόν όλα αυτά στο όριο, στην οροφή που έχουμε θέσει ως κανονιστικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει πραγματικά ανταγωνισμός δηλαδή. Για τις τιμές τώρα περιαγωγής δεδομένων, οι στήλες που βλέπετε <clears throat> δείχνουν τις ε, μέσες τιμές λιανικής για την περιαγωγή δεδομένων και στο τέλος έχετε την τιμή της ε, περιαγωγής χονδρικής. Βλέπετε λοιπόν ποιο είναι το κόστος όταν είσαστε σε μία σε περιαγωγή ε, που δεν ανήκει στον ίδιο με αυτή την ε, επιχείρηση η οποία είναι ο παροχός σας. Φτάνει λοιπόν τα 2 ευρώ ανά megabyte η τιμή των, ε, της περιαγωγής. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, ένα τεράστιο περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει μάλιστα διευρυνθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών που, δούμε, που βλέπουμε στην αγορά, θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλες λύσεις και όχι απλώς το να υπάρχει ένα ανώτατο όριο στις τιμές της περιαγωγής όπως είχαμε θεσπίσει το 2007. Αυτό ήταν απαραίτητο βέβαια να υπάρχει στον κανονισμό που είχε ζητηθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να εξετάσει και εναλλακτικέ ρυθμίσει, όχι μονάχα τη ρύθμιση ανωτά των ορίων τιμών, να δει αν υπάρχουν δυνατότητε να προωθήσουμε την αγορά περιαγωγή και την χρήση υποκαταστάτων στην αγορά του ρόμιν. Έχουμε λοιπόν καταλήξει σε μία νέα υβριδική, όπως τη λέμε, προσέγγιση, το πιο σημαντικό στην αγορά περιαγωγή σε μακροπρόθεσμη προοπτική είναι τα δομικά στοιχεία τα οποία θέλουμε να προτείνουμε στην ε, πρόταση της Κομισιόν. Αυτά τα διαφορετικά λοιπόν στοιχεία θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια έχουν σαν στόχο να διευρύνουν το πλαίσιο επιλογών του καταναλωτή ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των τιμών της περιαγωγής, μεγαλύτερη διαφάνεια για τον καταναλωτή όταν θέλει να επιλέξει τον πάροχο κινητών τηλεφωνικών υπηρεσιών. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνουν τους νέους πάροχους υπηρεσιών roaming να μπουν στην αγορά εάν το επιθυμούν. Εδώ βέβαια μπαίνουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες στο σύστημα, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα αυτά για τον λόγο αυτό χρειάζεται παραλύλο να διατηρήσουμε το σύστημα των οροφών για τις τιμές περιαγωγών, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα μέχρι ότου οι νέες διαρθρωτικές λύσεις γίνουν αποτελεσματικές. Να εξηγήσω λίγο περισσότερο τι είναι αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν. Υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Καταρχήν, υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι εύκολα στην ε, εφαρμογή τους και μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόλις εγκριθεί η νέα, ο νέος κανονισμός. Ο στόχος είναι <clears throat> να υπάρξει περαιτέρω πρόσβαση στην αγορά στους ε, κατόχους λεγόμενων εικονικών δικτύων κοινικής τηλεφωνίας, δηλαδή αυτών που δεν έχουν ένα δίκτυο με υποδομή δικό τους, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν λοιπόν την υποδομή που βρίσκεται με λογικούς όρους και θεωρούμε ότι μήνες, εάν υπάρχει μια λογική αίτηση και αν συμμορφώνεται με όλες τις προϋποθέσεις που έχουμε θεσπίσει μέσα σε δύο μήνες αυτή η εικονική υπάροχη υπηρεσιών κινητή τηλεφωνία θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υποδομή και να δίνουν υπηρεσίε στου χρήστε. Ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο ίσω είναι ακόμα πιο σημαντικό, να υπάρξουν οι δυνατότητες από τα μέσα του 2014 ο τελικός χρήστης να διαλέγει τον ε, πάροχο υπηρεσιών ε, περιαγωγής χωριστά από τον κανονικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, αν είσαστε ικανοποιημένος με τις υπηρεσίες που σας δίνει ο πάροχος υπηρεσιών στη χώρα σας, αλλά θέλετε να διαλέξετε τον πάροχο περιαγωγής όταν είστε σε μια άλλη χώρα, θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε τις τιμές και τις προσφορές των παρόχων υπηρεσίας και αν το βρείτε αυτό το πράγμα μπορείτε να κρατάτε τον δικό σας πάροχο στην χώρα που μένετε και να έχετε ένα χωριστό πάροχο για τις υπηρεσίες περιαγωγών για άλλες χώρες. Έτσι μπορεί ο καταναλωτής να διαλέγει με ένα φιλικό προς τον καταναλωτή και εύκολο τρόπο. Όπως σας είπα, αυτό θα χρειαστεί χρόνο, χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών. Θα πρέπει να δεχτούν κοινά πρότυπα, κοινές ε, αρχές για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα Στον κανονισμό αυτό είχαμε το όριο αποκοπής για την περιαγωγή, αλλά δεν εφαρμόστηκε αμέσως. Δόθηκε περίπου ένας χρόνος στους παρόχους για να εφαρμόσουν αυτή τη ρήτρα σε συνεργασία με, την, ε, με τους Ευρωπαίους ρυθμιστές. Μία αντίστοιχη προσέγγιση είναι αυτή που προτείνουμε εδώ πέρα με το να είναι χωριστό το τμήμα το οποίο αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγών. Σε δύο χρόνια λοιπόν αν εγκριθεί ο νέος κανονισμός, αν εγκριθεί στο τέλος του Ιουνίου 2012, σε δύο χρόνια από τότε, το, στο μέσο του 2014, θα υπάρχει δυνατότητα για τους καταναλωτές να διαλέγουν αυτόνομα τον πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής. Ενδιάμεσα όμως θα πρέπει να διατηρήσουμε την, το άνω όριο τιμών. <clears throat> Προτείνουμε λοιπόν να διατηρηθεί αυτό το άνω όριο τιμών μέχρι το 2016, αλλά το 2015 θα κάνουμε μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς, μια ανάλυση των καταστάσεων αγοράς και να ελέγξουμε το κατά πόσον αληθεύει και ευσταθεί η ιδέα ότι μπορεί η αγορά να λειτουργεί μετά από το 2016 χωρίς άνω όριο στο τίμημα της περιαγωγής. Τέλος, για την περιαγωγή δεδομένων που είναι το μόνο τμήμα το οποίο αυτή τη στιγμή σε λιανικό επίπεδο δεν καλύπτεται από ρυθμίσει. Βλέποντας ότι υπήρξαν μεν μειώσεις στην τιμή χονδρικής περιαγωγή δεδομένων, αλλά δεν είχαν καμία αντίκτυπο στι τιμές λιανικής για, τα, για την περιαγωγή δεδομένων, θα πρέπει να δούμε και εκεί πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα υψηλά περιθώρια. Όπως είδατε, είναι πάνω από 1 ευρώ ανά μεγαμπάιτ η τρέχουσα τιμή. Επομένως, ο στόχος μας είναι από το 2, να ξεκινήσουμε με ένα ανώτατο όριο που θα είναι 0,90 cents και θα μειωθεί αυτό το όριο στα 50 cents το 2014 για τη λιανική περιαγωγή δεδομένων. Όταν βλέπει κανείς αυτές τις προτάσεις, αν δει κανείς μονάχα τις τιμές και το κόστος, μπορεί να θεωρεί κανείς ότι εξακολουθούν να είναι μεγάλα τα περιθώρια κέρδους, η διαφορά μεταξύ τιμής χονδρικής και ελληνική και ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί εδώ. Αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα δύο στοιχεία, τα διαφορετικά μέτρα, τις διαφορετικέ λύσεις που προτείνουμε και το χάσμα, το περιθώριο κέρδους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα για να μπουν νέοι υπάροχοι υπηρεσιών στην αγορά. Επομένως, παρά το γεγονός ότι εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από αυξήσεις τιμών, δεν μπορούμε να συμπιέσουμε τις τιμές υπερβολικά προς τα κάτω, γιατί αυτό δεν θα δώσει κίνητρα σε νέους παρόχους να μπουν στην αγορά και να ανταγωνιστούν. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συνυπολογίσουμε και τα δύο στοιχεία όταν θέλουμε να εξετάσουμε την, όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε μάλλον την πρόταση αυτή της Κομισιόν και νομίζω ότι εδώ μπορώ να κλείσω την παρουσίαση μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαντελίν, να παρουσιάσουμε και την πιο πρόσφατη νομοθετική πρόταση και να έχουμε και τη γενική επισκόπηση προφανώ, Εάν θέλετε να θέσετε κάποια ερωτήματα, είμαστε στη διάθεσή σα για να απαντήσουμε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση αυτή η οποία προτείνεται, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι είναι καλό να ε, έχουμε και ένα κείμενο της ομιλίας σας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά προβλήματα που αναφέρατε για την περιαγωγή. Ίσως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Έρχομαι τώρα στους ομιλητές και ξεκινώ με τον κύριο Ρίμπιχ. Σας ευχαριστώ λέει κύριο Ρίμπιχ και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για τον κανονισμό περιαγωγή 3 που παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορίες. Και το ερώτημα πραγματικά είναι αν μπορούμε χωρίς αυτό το τεράστιο χάσμα τιμών χονδρικής λιανικής το οποίο αναφέρατε που μπορεί να φτάσει τιμή το χάσμα στο 1 ευρώ ανά megabyte είδα ότι σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης ζητάει κάποιος 13,9 ευρώ το megabyte. Λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε ένα ευρώ το μεγαμπάιτ μονάχα σαν χάσμα μεταξύ χονδρικής και λιανικής, γιατί πρέπει να πληρώνεις καταναλωτής τόσο πολύ πάνω από 10 ευρώ το μεγαμπάιτ σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ήδη σε πολλές χώρες ε, <clears throat> πακέτα που με 8 ευρώ παραγωγής χάρη έχει κανείς 8 γιγαμπάιτ πληροφοριών. Δηλαδή ένα γιγαμπάιτ που είναι 1000 μεγαμπάιτ δίνει, δίνεται με ένα ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ένα τεράστιο χάσμα τιμών. Αλλά εάν γυρίσει κανείς πάλι στο παράδειγμα που σας έδωσα προηγουμένως, αν θέλει κανείς να δουλέψει με ένα smartphone θα πληρώσει 13.000 παραπάνω για ένα gigabyte. Λοιπόν, 13.900 ευρώ έναντι 1 ευρώ στη χώρα που είναι κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ε, gigabyte και βγαίνει κανείς, πηγαίνει ξέρω εγώ έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι χιλιάδες παραπάνω. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσε να υπάρξει και ένα πιο ομοιόμορφο πλαίσιο για την ε, δημιουργία των τιμών αυτών και αν θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό. Και επίσης για τις τιμές στον τελικό καταναλωτή. Ο καθορισμός των τιμών στον τελικό καταναλωτή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτέλεσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Αν δεν είναι σαφές λοιπόν το ποιο είναι το πλαίσιο για τον καταναλωτή, αυτό θα δυσκολέψει και τη δημιουργία επενδύσεων και θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα χρήματα για επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ξέρουμε ότι οι εταιρείε κάνουν επενδύσεις μονάχα όταν έχουν κάποια εξασφάλιση ότι θα μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα κέρδη. Δεν πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε μονάχα για μέσα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για λογικό κέρδος ή για καταχρηστικό κέρδος και για πολλούς ε, στην κοινή γνώμη η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών εταιριών στον τομέα της περιαγωγής είναι καθαρά καταχρηστική για το 2016. Νομίζω ότι προχωράει τόσο γρήγορα η αγορά που ίσως θα πρέπει να θέσουμε πιο σύντομα χρονικά όρια, να μην περιμένουμε πέντε χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σε τρία-τέσσερα χρόνια με την τηλεφωνία τρι... τέταρτη γενιά θα υπάρχουν και νέε δυνατότητε, τι οποίε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και να λάβουμε υπόψη μα στη νέα αυτή κατάσταση. Κύριο Σοντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή για τις παρουσιάσεις. Υπό τη δικιά σας Γενική Διεύθυνση, θα ήθελα να μας ενημερώσετε για την αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Γιατί ήμουν εισηγητής για την αναθεώρηση αυτή και είχαμε κάπως ότι οι πυρογνώμονες δούλεψαν καλά, αλλά ότι η Επιτροπή άρχισε πάρα πολύ να παρουσιάσει την ανακοίνωσή της. Εγώ είχα 15 μέρες να κάνω την έκθεσή μου, πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή. Εμείς, η Επιτροπή μας δηλαδή εδώ, έπρεπε να κάνει τη δουλειά αυτή σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να μεταφέρει το δικό του μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ετοιμαστούν οι ε, προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για τις περιόδους 2011, 12 και 2013, όπου έχουμε 30 δις ευρώ να δαπανίσουμε συνολικά και πρόκειται για χρονιές, ε, θα έλεγα, εύθραυστες μια που δεν υπάρχει πραγματικά ανάκαμψη, αλλά δεν υπάρχει βέβαια και ε, καταστροφή. Συνεπώς, ρωτάω πρώτον, εσείς είσαστε ενήμερος και λάβατε υπόψη σας την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου μεταφέραμε τα μηνύματά μας και λέγαμε να απλοποιήσετε αυτές τις προσκλήσεις, διότι οι χρήστες θεωρούν ότι οι προποθέσει διατυπώνονται πάρα πολύ περίπλοκα. Έπειτα, το μήνυμα που λέει ότι πρέπει να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία κτλ. Στις προσκλήσεις αυτές ε, που εσείς ετοιμάσατε για τον Ιούλιο του 2011, 7,5 δις, αν δεν απατώμε για τη δικιά σας τη διεύθυνση, μπορείτε να μας πείτε λοιπόν περισσότερα γι' αυτό. Και όσον αφορά τώρα το, την περιαγωγή για την μείωση των τιμών σε αυτό. Οι πολίτες μας είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές και πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε λοιπόν εσείς να μας διασφαλίσετε ότι σε συμφωνία με τους ρυθμιστές που ασχολούνται με τον καθορισμό των τιμών της υποδομής, η μείωση αυτή των τιμών δεν θα επηρεάσει και τις επενδύσεις στα δίκτυα έτσι ώστε να υπάρχει κάλυψη σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και να υπάρχει και ανανέωση των δικτύων, ε, σύμφωνα που να συνάδει δηλαδή με τις τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί υπάρχουν εξελίξεις για πολύ μεγάλη ροή, δυναμικό, και οι πολίτες μερικές φορές έχουν την αίσθηση σε κάποια σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν βρίσκονται επίση όρις με τους υπόλοιπους. Δεν έχουν δηλαδή τις κατάλληλες υποδομές για να έχουν εξίσου πρόσβαση στα δίκτυα. Έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι η δικιά σα συλλογική είναι πολύ αστική. Δηλαδή θεωρείτε, ωραία, στι πόλει έχουμε πολλού πελάτε, οπότε το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι η μείωση των τιμών. Ναι, αλλά μείωση των τιμών σημαίνει ότι οι φορεί έχουν λιγότερα χρήματα και άρα επενδύουν και λιγότερο. Εσεί μπορείτε να μα εγγυηθείτε ότι οι επενδύσει θα συνεχίσουν, θα είναι παρούσε και ότι όλοι οι πολίτε θα έχουν πρόσβαση στι υπηρεσίε αυτέ όπου και αν βρίσκονται στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάδελφος όχι αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη νέα πρόταση που υπάρχει όσον αφορά την περιαγωγή, το roaming. Νομίζω ότι έχουμε μια αγορά που δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό ο κανονισμός αυτός να βελτιωθεί, η ρύθμιση αυτή να βελτιωθεί, να βελτιωθεί δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Η ερώτησή μου είναι εξή. Έχετε προβλέψει, μια που με διάφορες τροπολογίες προσπαθούμε εμείς να βελτιώσουμε το κείμενο, έχετε προβλέψει τα εξή. Πρώτον, πιστεύουμε ότι δεν έχει λυθεί το θέμα των συνόρων, των κρατών μελών δηλαδή, με άλλες χώρες. Και το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί, οι παρεμβολές. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα σε μια χώρα μέλος οι επικοινωνίες σε διασυνοριακές περιοχές να παρεμβαίνει η περιαγωγή από τις γειτονικέ χώρες για τα SMS, για τα μηνύματα, για την μεταβίβαση δεδομένων. Έτσι, ο λογαριασμός που παίρνουν οι καταναλωτές στις διασυνοριακές περιοχές είναι πάρα πολύ ψηλός. Αυτό θα πρέπει να λυθεί. Και το δεύτερο, το οποίο θέλω να σας αναφέρω, είναι το εξής. Πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει ότι για το θέμα της περιαγωγής τα SMS, τα γραπτά μηνύματα δηλαδή, καθυστερούν. Μερικές φορές περνάνε και μέρες μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ θα έπρεπε να μπουν κάποια κριτήρια ε, επιδόσεων. Έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες καθυστερήσεις. Να, γιατί ο ρόλος που έχει ένα τέτοιο μήνυμα ή αποστολή ενό τέτοιου μηνύματο είναι να φτάνει άμεσα στον προορισμό του, όπω ε, όταν παίρνουμε τηλέφωνο δηλαδή. Να μην καθυστερεί. Κάτι άλλο που θέλω να θίξω εδώ είναι το θέμα των νομοθετικών πρωτοβουλειών που θα αναλυθούν στο μέλλον για την ηλεκτρονική ταυτότητα και για την ηλεκτρονική υπογραφή. Εμείς ε, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δύο αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναγγελθεί. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι από του χρόνου θα δουλέψει πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Ελπίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάτι θεμελιώδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Καβάλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Γενικό Διευθυντή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το νέο ταμείο. Για τις διευκολύνσεις υποδομών στην διασύνδεση μέσα στην Ευρώπη. Για τις προτεραιότητες, δηλαδή που τίθενται και τα καταπροτεραιότητα προγράμματα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή, φαντάζομαι ότι εδώ θα για διάφορες χώρες. Βλέπετε, έχουμε μια εμπειρία από το παρελθόν πολύ χαμηλών επιδόσεων των προγραμμάτων που έχουν να κάνουν αυτά τα θέματα. Ιδιαίτερα στη χώρα μου, το θέμα της οικονομικής ανά, ε, ανάκαμψης, το θέμα των πληροφοριών, το θέμα της ευρυζωνικότητας, είναι πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν καλά στη χώρα μου. Η εφαρμογή τους δηλαδή καθυστερεί πάρα πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουν σαφείς και εύκολα κατανοητοί κανόνες. Υπάρχει και ένα θέμα με την συγχρηματοδότηση, γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η συγχρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή λάβατε υπόψη σας ε, το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι αυτό ήταν ε, το πρόβλημα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή το γεγονός ότι έπρεπε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στα δίκτυα και να τους ε, βοηθήσουμε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με τα δίκτυα. Αυτό απέτυχε στο παρελθόν, τουλάχιστον από πλευρά του Κοινοβουλίου, δεν εγκρίθηκε. Επομένως, ρωτώ, αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την είσοδο στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την είσοδό τους στα δίκτυα, διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις τους εμποδίζουν να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο. Η κυρία Ριέρα Μαρντουέλ έχει το λόγο. Α, συγγνώμη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, συγγνώμη. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα, αλλά και εσάς για την παρουσία σας εδώ και τους δυο σας λοιπόν για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Όπως είπατε είναι μια πολύ καλή στιγμή αυτή για να δούμε τι μας περιμένει το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Νομίζω ότι ανατρέξατε πάρα πολύ καλά στα διάφορα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε, μεταξύ άλλων την περιαγωγή, το roaming, Όλα αυτά τα θέματα είναι ζητήματα για τα οποία θα συζητήσουμε πολύ τους επόμενους μήνες. Θέλω να προσθέσω όμως μερικές ερωτήσεις στον κατάλογο, που έτσι είναι αρκετά πλήρης. Παρ' όλα αυτά έχω να προσθέσω κάποια πράγματα, γιατί όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα μου υπέβαλε πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012. Από αυτού λοιπόν έχω να σχολιάσω τρία θέματα που αναφέρονται στην πρότασή μας και για τα οποία θέλουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της δικιάς σας Γενικής Διεύθυνσης. Πρώτον, είναι το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και ιδιαίτερα το θέμα της δαφικότητας σε τρεις δράσεις. Συμφωνούμε για το ότι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς ε, απαιτεί συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική υπογραφή, προσφορές ηλεκτρονικά και άλλα πράγματα στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Όμως, προκειμένου να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών και να υπάρχει δραστηριότητα διασυνοριακά επίσης ώρες, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την βιωσιμότητα της αρχής αυτής της αδερφικότητας. Και για να τα πω σύντομα, θέλω να αναφερθώ στο εξής. Επίγεινε, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο σταθερό, να ξαναδούμε το ήδη υπάρχουν για τις τηλεπικοινωνίες και να φροντίσουμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις για το θέμα της ταχύτητας, ε, σύνδεσης και άλλα σχετικά θέματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νομική ασφάλεια και μια καλή τιμή για τον χρήστη, για τον καταναλωτή. Τέλος, εν ώψη του μελλοντικού προγράμματος πλαισίου, θα θέλαμε και εμείς να δούμε αύξηση της χρηματοδότησης για την πληροφορική. Εμείς το στηρίζουμε στην ομάδα μας γι' αυτό. Και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αναδυόμενων αγορών όπως είναι αυτές που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία στον τομέα της υγείας, με τις οικολογικές μεταφορές ή άλλες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τα ευφύ δίκτυα ενέργειας, αλλά και άλλα που αναφέρθηκαν εδώ. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Μαντελίν. Το πιο ενδιαφέρον στη νέα σας πρόταση είναι τώρα οι νέες δομές που έχετε προτείνει. Γιατί όμως δεν θέλετε να προχωρήσουμε πιο, με πιο γρήγορα βήματα. Γιατί πρέπει να περιμένουμε το 2016, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει να συνεχίσουμε με τα, όρια των, τα ανώτατα όρια των τιμών. Αυτό δεν μου άρεσε ποτέ λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα εφαρμοστεί το νέο σύστημα αυτό, το ταχύτερο. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, πολύ και για τα σχόλια και τις ερωτήσεις και για τα μηνύματα αν θέλετε τα πολύ ενδιαφέροντα να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις που δεν αφορούν το roaming την, ε, και την περιαγωγή και μετά ε, να ομαδοποιήσουμε τις υπόλοιπες. Λοιπόν, για τον κύριο Οντί, για την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου. όλα αυτά είχαν χωνευθεί, αν θέλετε, πριν ξεκινήσω εγώ. Όμως, υπό την ηγεσία της κυρίας Γκέγγεν Γουίνς είχαν γίνει πολύ συγκεκριμένες ε, προτάσεις για απλούστευση που όμως ε, δεν έγιναν ε, με τον ενθουσιασμό που θα περιμέναμε δεκτές οι προτάσεις αυτές από πολλούς εδώ σε αυτό εδώ το, το, όργανο και Προφανώς πολλοί συνάδελφοι καταλαβαίνουν ε, γιατί δεν είναι καθόλου ε, ικανοποιημένες ε, οι μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι στην Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, στις υπηρεσίες ελέγχου, έχουμε την υποστήριξη των συναδέλφων για να προχωρήσουμε για απλούστευση και στο πολιετές πρόγραμμα ε, χρηματοδότησης και με ορίζοντα το 2020 ε, Υπάρχουν ιδέες οι οποίες αξιολογούνται στην Κομισιό Έχουμε την διευκόλυνση στο Ταμείο το ΦΕΤΑ και προσπαθούμε εκεί να κάνουμε ό,τι δυνατόν μπορούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, κάναμε όλα όσα οι αναθεωρητές, αν θέλετε, ε, περίμεναν από εμά. Όχι βέβαια. Κάποιες προτάσεις χαθήκανε κάπου στο δρόμο και στην Κομισιόν και εδώ. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση στην την, ε, την ε, ηλεκτρονική ταυτότητα και την ηλεκτρονική υπογραφή, το φθινόπωρο θα έχουμε μια συλλογική απάντηση και όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική ταυτότητα και την ηλεκτρονική υπογραφή. Γιατί η ηλεκτρονική υπογραφή χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Είχαμε μια καλή απάντηση αν θέλετε από τα πιλωτικά προγράμματα που κάναμε. Τώρα θέλουμε να συνδυάσουμε και, τα δύο, και τις δύο προτάσεις και για την ηλεκτρονική ταυτότητα και την ηλεκτρονική υπογραφή γιατί θεωρούμε ότι και τα δύο αυτά θέματα συνδέονται. Τώρα, για το θέμα που έθεσε η κυρία Τικάου επίσης ε, για τις ε, μεθοριακές περιοχές. Μία λύση είναι να έχει την δυνατότητα, γιατί τα περισσότερα ούτως ή άλλως τηλέφωνα το ε, ε, επιτρέπουν, να επιλέξεις τον δικό σου τον τοπικό φορέα και όταν είσαι στην, στην περιοχή σου και μονάχα όταν απομακρυνθείς να έχει το γενικό roaming. Τώρα οι παρεμβολές και στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πολλές φορές όντως χρειάζεται λίγος χρόνος όσον αφορά δηλαδή την αποστολή των μηνυμάτων. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί, δεν άπτεται όμως άμεσα της περιαγωγής. Κυρία Καβάριο μίλησε για την Ένωση στην Ευρώπη. Σε αυτό το στάδιο έχουμε φτάσει στις υπηρεσίες ε, της Κομισιόν σε μια γενικότερη αποδοχή και έχουμε υποβάλει μια πρόταση για το γενικό ποσό το οποίο θέλουμε να ξοδέψουμε. Τώρα για συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να γίνει μια κατανομή αν θέλετε ανάμεσα στην ενέργεια της ε, μεταφορές και της τηλεπικοινωνίες. Εμείς ε, θεωρούμε ότι οι επικοινωνίες είναι το μικρότερο, ο μικρότερος τομέας από τους υπόλοιπους δύο όσον αφορά τις οικονομικές ανάγκες. Για το πώς τώρα θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά πρέπει να ξέρετε ότι από το ε, πρόγραμμα ανόρθωσης έχουμε διδαχθεί κάποια πράγματα. Παραδείγματο χάρη, θα πρέπει... Δεν μπορεί, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ανάπτυξη της υπαίθρου να τους αναθέτουμε χρήματα για να εφαρμόσουν ευρυζωνικά προγράμματα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον οικονομικό επίπεδο, στην, ε, σε τράπεζες. Τώρα, όσον αφορά την συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να βρούμε κάποιες καινοτόμες λύσεις, να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τους πόρους που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και να ξεπεράσουμε τα κάποια κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις πηγές χρηματοδότησης, είτε είναι αυτά διαδροτικά ταμεία, είτε εθνική πόρη, είτε κοινοτική πόρη κτλ η ιδιωτική πόροι. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Μαντούρο. Καταρχάς, ε, καλωσορίζουμε την υποστήριξή σας γιατί τη χρειαζόμαστε. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ε, αρμόδιοι επίτροποι, η κυρία Κρούς και ο κύριος Μπαχνιέ ε, συνεργάζονται μαζί μας ή εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε όμως χρειαζόμαστε να γίνει μια έρευνα για το κόστος της μη ύπαρξης της Ευρώπης στον τομέα αυτό και ελπίζουμε ότι από αυτή την έκθεση θα έχουμε τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση σε εδαφικό επίπεδο. Τώρα για την νομική βεβαιότητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επανέρχομαι στα προηγούμενα σχόλια που έγιναν. Τώρα ξεκινήσουμε, τα πρώτα μας βήματα ε, Βέβαια, για το τρίτο πακέτο ακόμα υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή της απαραίτητης νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και προφανώς δεν έχουμε ένα σταθερό και ασφαλές νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Γιατί χρειαζόμαστε και καλύτερη, για να, το, οποίο, το οποίο χρειαζόμαστε για να έχουμε και μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή. Τώρα, για την καινοτομία και την έρευνα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι πυλώνες δραστηριοτήτων. Το ένα είναι οι επικοινωνίες και ε, που θα λάβει υπόψη ε, την, ε, έξυπνη έρευνα, την έξυπνη ενέργεια, την πρόοδο κτλ. Και ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις τεχνολογίες και αυτόν τον πυλώνα δεν πρέπει να το χάσουμε από το ε, μυαλό μας. Διότι καλά να μιλάμε στον αδελφό μας, την ξαδέλφη μας, την πεθερά μας για τις ε, προκλήσεις, όμως οι προκλήσεις ε, αφορούν τους ειδικού για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιες, κάποια προηγμένη, προηγμένη τεχνολογία. Τώρα, για την περιαγωγή θα απαντήσω στην ερώτηση του κύριου Ρούμπιχ και του Προέδρου. Η Επιτροπή είναι εγωκεντρική. Δηλαδή από τη στιγμή που αποφασίσουμε τι θέλουμε να προτείνουμε, όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε τόσο καλύτερα. Και θέλουμε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό που θα, είναι, θα προσεγγίσουν τον περισσότερο την δική μας πρόταση. Τώρα, για είναι περίοδο, τη μεταβατική περίοδο. Αυτό το είναι ένα πιο ευαίσθητο θέμα για τον έλεγχο, για ε, τις στη τιμές ε, και για το roaming. Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν την ίδια στιγμή που αποφασίσει ο νομοθέτης με μια ελάχιστη περίοδο μεταφοράς, ε, μεταβατική περίοδο για να σεβαστούμε τα υπάρχοντα συμβόλαια. Όμως όσον αφορά τις διαρθρωτικές λύσεις πρέπει να αλλάξει η αγορά ίδια. Δηλαδή, οι διαρθρωτικές λύσεις τι σημαίνουν ότι κάθε φορά που ένας πελάτης μπαίνει σε ένα μαγαζί και υπογράφει ένα νέο συμβόλαιο ή κάθε φορά που παίρνουν τις λεπτομέρειες ε, του λογαριασμού τους, θα πρέπει να θέτει το ερώτημα έχω κάνει τη σωστή συμφωνία. Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ξέρουν ποιο είναι το κόστος της περιαγωγής στο ισχύον του συμβόλαιο ή το, το συμβόλαιο που τους προτείνει ο φορέας τους, ο προμηθευτής τους, αλλά θα πρέπει να ξέρουν και τους όρους των άλλων εταιριών. Και δεν ξέρω εάν η αγορά μπορεί να προσφέρει αυτού του είδους πληροφορίες. Άρα εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε τον πιο γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο ε, τόσο, τόσο γρήγορα έτσι ώστε να μην ε, ε, έχει ο καταναλωτής τις πληροφορίες που χρειάζεται. Εγκαίρος. Τώρα, η ερώτηση που έκανε και ο κύριος Οντί και ο κύριος Ρούμπιχ για την βιωσιμότητα του προτινόμενου μοντέλου. Σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε προτείνει και εμείς και η κυρία Κρούς, είναι ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με μεγάλες ταχύτητες σε ευρυζωνικές ζώνες στην Ευρώπη. Ε, και πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας αυτό. Ε, και ο πρόεδρος Μπαρόζο και άλλοι ε, εκπρόσωποι της Κομισιό ασχολούνται με το θέμα αυτό αυτές τις μέρες. Και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί μια απόφαση ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, και να προσπαθήσουμε περισσότερο στο θέμα. Αυτή η περαιτέρω προσπάθεια δεν σημαίνει όμως ότι η αγορά θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Ε, δεν υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στα περιθώρια κέρδους ε, για τις, για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αφενός και τις επενδύσεις αφετέρου. Δεν υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στα δύο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου εμείς πιστεύουμε, όπως δείχνουν και οι διαφάνειες, ότι υπάρχει πολύ περιθώριο να... Ε, πολύ μεγάλο περιθώριο όσον αφορά την μείωση των τιμών για τη μεταφορά δεδομένων και την, ε, χωρίς να περιορίσουμε τις επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή που αυτό που μετράει είναι όγκος. Στη Δανία, ας πούμε, το 90% ε, των, ε, γυναικο, των νοικοκυριών έχουν ε, ευρυζωνική ε, επικοινωνία από τα σπίτια τους, όμως θέλουν πολύ φτηνά συμβόλαια. Αυτό τους μετράει. Αυτό του μετράει για αυτούς. Γιατί ακριβώς δεν έχει προσθεθεί ακόμα το περιεχόμενο. Και εδώ επανέλθουμε στο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη είναι να δημιουργήσουμε πιο ενδιαφέρουσα αγορά για ένα σεξι αν θέλετε περιεχόμενο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Και μετά μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις ε, υπόλοιπες προκλήσεις. Τώρα, για τα μηνύματα, το κατά πόσον το... Συμφωνώ ότι το μήνυμα ανεξάρτητα από το αν είναι περιαγωγής ε, ή είναι ένα μήνυμα που λέει ότι θα έρθω, θα αργήσω λίγο να επιστρέψω στο σπίτι μου, στο σπίτι, ε, είναι όντως ανησυχητικό εάν φτάνει μετά από πολλές ώρες. Και εκεί θα πρέπει να το δούμε. Τώρα για την ερώτηση του κυρίου Ράμστορφ και εδώ ολοκληρώνω τι απαντήσει μου. Αυτό αυτή η πρόταση που έκανε ο Βάζα προηγουμένως συμφωνούμε από ότι από σήμερα είναι ε, εφικτό για τους τοπικούς, τοπικές εταιρείες να επιτρέψουν την πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα. Σε μικρομεσαίους providers δηλαδή. Θέλουμε αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ένα δίκτυο σε μια χώρα να συνάπτουν ε, συμφωνίες με όλους όσους το επιθυμούν. Άρα θέλουμε να βελτιώσουμε την δυνατότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μια σφαιρική κάλυψη στην Ευρώπη των 27. Εάν και εφόσον το πετύχουμε αυτό, τότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε μια διαρθρωτική λύση. Τώρα, έχουμε προχωρήσει αρκετά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε, αυτή, να επιβάλλουμε μάλλον αυτή την υποχρέωση. Αυτό θα το αποφασίσει ο νομοθέτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εξ ονόματος όλων μπορώ να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του κύριο Μαντελίν για την παρουσίασή του και τις απαντήσεις που μας έδωσε, για τις πλήρες πληροφορίες που μας έδωσε, για τις εξηγήσει που μας παρέσχε. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τις μεταγενέστερες συζητήσεις μας. Τις επόμενες εβδομάδες, ίσως όχι εβδομάδες, στους επόμενους μήνες πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε σε επαφή για να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Thank you, λέει ο Πρόεδρος.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 Okay, Πάμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Okay, we Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε αν δουλεύουν τα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Αν συμφωνείτε, ποτού προχωρήσουμε στην, ε, στην πραγματική ψηφοφορία. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία με το ερώτημα ναι ή όχι. <laughs> Διακόπτουμε τις συνεδρίες, κλείνουμε τις συνεδρίες και πάμε όλοι διακοπές. Λοιπόν, ψηφίστε ή ναι ή όχι για αυτή την πρόταση. Okay, vote is closed. Πέρας προφορίες. Oh. Δεν με εκπλήττει το αποτέλεσμα. 23 ψήφοι υπέρ. Εντάξει. 6 κατά, Εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την κανονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε πρώτα. Έκθεση της κυρίας Βίκη Φόρτ. Ασφάλεια ε, εξορίξεων φυσικού αερίου και πετρελαίου που γίνεται με υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Ξεκινάμε. Τροπολογία 31. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές δεκτή. 33. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 και 37 εκπίπτουμε, 34 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 και 40 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Πάμε στην... Ε, πάμε στην 40... 41. 41 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πορ. Απορ. Πάμε λίγο, πιο, πάμε λίγο γρήγορα ίσως. Μερικέ φορέ πρέπει να, να είμαστε προσεκτικοί με την αλληλουχία των τροπολογιών. 43 και πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ωραία, ευχαριστώ. 44, όχι εκπίπτει. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Απασχόληση 2. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Απασχόληση 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απασχόληση 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50, 57. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 59. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ Πρώτο τμήμα υπέρ Κατά αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα που ψηφίζει παραπάνω. Αυτό είναι νέο, νοφανές φαινόμενο, λέει ο πρόεδρος. Πριν από τις διακοπές, αυτό είναι εντυπωσιακό. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Όχι, όχι, το τρίτο τμήμα εκπίπτει. Εντάξει. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67, όχι 66 εκπίπτει. 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6α ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση 8 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Ε, κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απολύτω το δεύτερο τμήμα. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 77 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 90 ψήφι υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. εκπίπτουν εκπίπτουν 95 ψήφοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 και 14 του περιβάλλοντος με μια προφορική τροπολογία του εισαγητή. Είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 107 εκπίπτει, 103 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 και NV15 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 109. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 καθώς και NV20 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 130 Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτουν. Δεύτερο τμήμα της NV18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. NV18 το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Επαναλαμβάνω. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 σαν προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απασχόληση έμπλη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». 143 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλεπτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 7 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10... 13 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 19 υπέρ. Παρακαλώ. 19 υπέρ κατά και πάλι από την αρχή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 μήπως μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες οι μπούρμπουλες μέχρι την 30 όλες μαζί μέχρι την 30 ωραία 23 μέχρι 30 ψήφι όχι δεν μπορώ όχι για ποια δεν θέλετε να ψηφίσουμε μαζί. 23 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 1 ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή 2 και 4 που πάνε μαζί ταυτόσιμες ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτές 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτές δεκτή 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Εμπλένα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εμπλέξη υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εμ10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εμπλ12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εμπλ16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 όχι 21 έχει εκπέσει, 21 έμπλ υπέρ κατά αποχές δεκτή. NV1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. NV31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. NV36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτό είναι. Τελική ψηφοφορία λοιπόν <clears throat> με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. And... Closed. Πέρας. Πέρας. Σαφές αποτέλεσμα. 41-6. Συγχαρητήρια στην κυρία Φόρντ. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Δεν ήταν εύκολη ψηφοφορία, αλλά είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ήταν το αποτέλεσμα όχι μονάχα πολλών ψηφοφοριών, αλλά και πολύ δύσκολη συνεννόησης με άλλες ε, επιτροπές. Κύριε Φόρ, θέλετε να πείτε κάτι. Λέω απλώ ευχαριστώ στου συναδέλφου μου από τι άλλε πολιτικέ ομάδε, γιατί όπω είδατε στον κατάλογο ψηφοφοριών εργαστήκαμε πάρα πολύ, ακόμα και πριν φτάσουμε την προθεσμία για τι τροπολογίε, για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιε συμβαστικέ λύσει. Σα ευχαριστώ λοιπόν τα μάλα, όλα τα μέλη των άλλων πολιτικών ομάδων που συνεργαστήκαν μαζί μου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ναι, ναι, χειροκροτήστε όλοι. Είναι πολύ σωστό. Ερχόμαστε στην έκθεση Μαρκάκη για τη διαφάνεια της αγοράς ενεργείας και την ακαιρεότητά της. Υπάρχει ένα συμβαστικό κείμενο. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, κατευθείαν ηλεκτρονικά. Με μία τροπολογία μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μία τροπολογία είναι πιο απλό. Ε? Ηλεκτρονικά με μία τροπολογία για τις τρεις αποφάσεις. Εντάξει. Closed. Πέρασε προφορίες. Όλα εντάξει. Συγχαρητήρια κύριε Χατζημαρκάκη. Και προχωρούμε τώρα στην επόμενη έκθεση, την έκθεση Σιμάνσκι. Ξεκινάμε με τη συμβαστική 1. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Όχι, όχι, όχι, λέει κάποιο. Έλεγχο για την 11, Όπω θέλετε. Βεβαίω. Πάμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται σαφώ. Ναι, ναι, είναι σαφές. Δεκατέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 15 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Α... Έλεγχος. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα, ηλεκτρονικός έλεγχος, αυτή την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26, 27 και 28 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 29. Θέλετε έλεγχο. 26 με 28. Ηλεκτρονικός έλεγχος αρχίζει. Ψηφοφορία. Πέρας. Στο τσίμα τσίμα. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Για την 29 θέλετε έλεγχο. Καλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Και απορρίπτεται με ισοψηφία. 30 ψήφι υπέρ. υπέρ. Κατά. Απόχε εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος στο πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Στη 40. 4-0. 4-0. Πρώτο τμήμα. Λήξεις. Και απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32 το δεύτερο τμήμα μονάχα ψήφι υπέρ. Το πρώτο τμήμα έχει εκπέσει. Κατά έλεγχος δεύτερο τμήμα της 32. Άρχεται. Ποιος? Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Εντάξει τώρα. Όχι. Κάποιος πρέπει να φύγει. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 ε- απορρίπτεται. Απορρίπτεται, ναι. Κάνουμε έλεγχο λοιπόν, εντάξει, την 39. Πάλι ένας περισσεύει από το ΕΛΚ. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 σε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα 41 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 42 υπέρ. Κατά Έλεγχος. Στη 42. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 την ψηφίζει ο πρώτος αλλά μάλλον εκπίπτει. Εκπίπτει. Εκπίπτει και η 46. Εκπίπτει. 47 έχει αποσυρθεί. 49. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Έλεγχος 49. Βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται όπως σας έλεγα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Ένα, σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιμάνσκι. Και αυτό έχει κλείσει αισίως. Ωραία. Τελευταία ψηφοφορία λοιπόν τώρα. Το ψήφισμα για την προφορική ερώτηση. Θα ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες αν συμφωνείτε. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το παγιωμένο ε, κείμενο, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται και αυτό. Και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο τμήμα της συνεδριασής μας. Τέλος οι ψηφοφορίες. Έχουμε τώρα την επίσκεψη του Πολωνού Υπουργού που δεν είναι εδώ παρόν όμως. Αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι δεν, θα έρθει μέχρι τις 11.30 ο κύριος ε, Υπουργός. Λέει η γραμματεία μάλλον στις 11.30 θα έρθει ο κύριος Υπουργός. Λοιπόν, διακόπτουμε μέχρι τις 11.30. Δεν έχει τώρα λόγο να χρονοτριβούμε. Πείτε καφέ, φτιάξτε τις βαλίτσες σας, κάντε ό,τι θεωρείτε σκόπιμο και πρόσφορο. Jesus.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

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και πάλι μετά από τη σύντομη διακοπή μας. Μπορούμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Παύλακ, τον ε, αντιπρόεδρο της πολωνικής κυβέρνησης που είναι ο υπεύθυνο υπουργό για οικονομικών. Αυτό είναι μεγάλη σημασία. Αυτή <clears throat> η παρουσία του χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ήδη από την αρχή της ε, πολωνικής προεδρίας Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα να μιλήσουμε και με τον κύριο Παύλακ και με άλλους εκπροσώπους της πολωνικής κυβέρνησης, γιατί βρισκόμαστε στην Πολωνία. Ήταν μια καταπληκτική επίσκεψη, πολύ καλά οργανωμένη, που μπόρεσαμε να συλλέξουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες όλοι αυτοί που ήμασταν παρόντες. Θα κλείσω λοιπόν εδώ πέρα αυτή την παρουσίαση και σας παρακαλώ κύριε Παύλακ να κάνετε την εισαγωγική σας ε, παρουσίαση και μετά οι συνάδελφοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Στις 12.30 βέβαια πρέπει να κλείσουμε, γιατί τελειώνει και το ωράριο των ε, ε, διερμηνέων που κάπως ξεπέρασαν τις, ε, το ωράριο της χθες το βράδυ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να έρθω και να σας δω. Χαίρομαι γιατί έτσι θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και με τη βιομηχανία. Ελπίζω η Πολωνική Προεδρία να αποδειχθεί μια καρποφόρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Προεδρία και για την Πολωνία. Γνωρίζω ότι άλλοι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο Υπουργός για την Επιστήμη και την Ανώτατη Εκπαίδευση, Κουτρίτσκα, ο κύριος Γκροβάτση επίσης θα έρθει και θα σας δει που είναι υπεύθυνο για τις υποδομές και ο κύριος Μίλλερ επίσης, ο οποίος εκπροσωπεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας στον τομέα της βιομηχανίας και της ενέργειας. Όσον αφορά την Πολωνική Προεδρία λοιπόν, προτείνουμε να επικεντρωθούμε σε τρεις τομείς. Αν δούμε δηλαδή συνολικά την ε, Πολωνική Προεδρία, το ένα θέμα είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τη βλέπουμε την ολοκλήρωση εμείς σαν πηγή ανάπτυξης. Η δεύτερη, ο δεύτερος τομέας μας είναι μια ασφαλής Ευρώπη ασφαλής διατροφή, δηλαδή ενέργεια, ασφάλεια προμήθειας δηλαδή. Και το άλλο είναι ωφέλη από μια Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο. Ο Υπουργό Οικονομικών είναι υπεύθυνο βέβαια για αυτά τα τρία ζητήματα. Έτσι σήμερα θα επικεντρωθούμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την βιομηχανία και την ενέργεια. Θα ξεκινήσω λοιπόν με λίγα λόγια όσον αφορά την πολιτική ενέργειας. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Εδώ θα αναφερθώ βέβαια στην εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε εμείς ότι το κυριότερο μέλημά μας είναι να έχουμε γερά θεμέλια στην εξωτερική διάσταση της ενεργειακής μας πολιτικής, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις χώρες που μας προμηθεύουν, που παράγουν ενέργεια και μας την προμηθεύουν, είναι ένα σημαντικός παράγοντας για μας και οι σχέσεις μας μαζί τους είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε όλος ιδιαίτερος. Είπαμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την εξωτερική διάσταση, γιατί έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα, πιστεύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διεθνή σκηνή και έτσι θα βελτιωθούν και οι προθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και οικονομής κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής τι σημαίνει. Σημαίνει για μας ότι πρέπει να έχουμε δύο μηχανισμούς, όπως λέει και το Συμβούλιο. Ο ένας είναι ο συντονισμός. Είναι ένας μηχανισμός δηλαδή, ο οποίος θα μας βοηθήσει να απλοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τις θέσει των κρατών μελών και των διαφόρων Ινστιτούτων που ασχολούνται με την ενέργεια. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η αλληλεγγύη. Έτσι θα διασφαλίσουμε ε, τις δυνατότητες που έχει κάθε χώρα και το κάθε Ινστιτούτο που ασχολείται με την ενέργεια για να λύνει ό,τι ε, προβλήματα προκύπτουν διμερώς ή όχι. Ένα άλλο θέμα πάνω στο οποίο θα επικεντρωθούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας για να ενισχύσουμε την εξωτερική αυτή διάσταση θα είναι η επέκταση του κοινοτικού κεκτημένου και σε άλλες χώρες. Θα επικεντρωθούμε στην επέκταση του κοινοτικού κεκτημένου στις γείτονες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα φροντίσουμε και για την επικύρωση της συνθήκης για την ενέργεια σε μια ευρεία κλίμακα χρησιμοποιώντας Θέλουμε δηλαδή να χρησιμοποιούν όλοι τους ίδιους μηχανισμούς, τα ίδια συστήματα, γιατί τότε θα είναι πιο εύκολο να συνομιλούμε με τους εταίρους μας. Και η εξωτερική μας πολιτική για την ενέργεια είναι κάτι που θα συζητηθεί στο Φράτσροφ το Σεπτέμβριο. Ο δεύτερος τομέας που έχει να κάνει με την ενέργεια και όπου θα επικεντρωθούμε είναι το θέμα της ασφάλειας προμήθειας ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και κατά την Προεδρία μας αυτό το θέμα και η σχετική οδηγία θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες μέχρι τώρα για να πετύχουμε το στόχο του 20% αύξησης της ασφάλειας προμήθειας στην ενέργεια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, μόνο το μισό θα πετύχει. Προκειμένου λοιπόν να πετύχουμε πλήρως την εφαρμογή του στόχου αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράσεις στον τομέα της μεταφοράς, ε, της οικοδόμησης ε, και του εξοπλισμού και η Πολωνική Προεδρία θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη προκειμένου να αναλάβουν τέτοιες δράσεις. Προτείνουμε λοιπόν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασιών όσον αφορά τη νέα οδηγία για την ασφάλεια προμήθειας. Η Πολωνική Προεδρία επιθυμεί το Σεπτέμβριο στη συνάντηση του Συμβουλίου να εγκριθεί μια έκθεση προόδου για την οδηγία αυτή. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα επικεντρωθεί η Προεδρία μας είναι νέα συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση το Energy Star. Κατά την Πολωνική Προεδρία θέλουμε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της νέας συμφωνίας με την Αμερική. Και κατά την Πολωνική Προεδρία επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο προτάσεις για επικύρωση της νέας συμφωνίας αλλά και σχέδιο που προετοιμάζει κανονισμό. Η Πολωνική Προεδρία θα αγωνιστεί προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στον τομέα αυτό. Στις 24 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου, θα ενημερώσουμε για την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό. Κάτι άλλο είναι οι ενεργειακές υποδομές. Και εδώ το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την οικοδόμηση υποδομών. Πολύ σημαντικό θέμα και για τους τρεις τομείς ενεργειακής μας πολιτικής η Πολωνική Προεδρία περιμένει τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο φθινόπωρο. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ο δικός χάρτης για την ενέργεια το 2050 που θα αναφέρεται βέβαια στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και με τις επιπτώσεις των δράσεων που αναλαμβάνονται για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γιατί έχουμε και τέρους με τους οποίους πρέπει να υπάρχει συμφωνία, αλλιώς δεν μπορούμε να πετύχουμε. Υπάρχει ενεργειακή πολιτική, υπάρχει επίσης η πολιτική για το περιβάλλον και η ευρωπαϊκή οικονομία που επηρεάζουν την κατάσταση. Ο άλλος τομέας που θα μας απασχολήσει είναι η ρύθμιση REMIT, κάτι στο οποίο θα επικεντρωθούμε γιατί ο κανονισμός αυτός θα μας βοηθήσει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή στις αγορές και θα συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι η ασφάλεια offshore όλων των εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου. Εδώ θέλουμε προδιαγραφές ε, ανώτατης ασφάλειας για να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους που απασχολούνται στον τομέα αυτών στην Ευρώπη. Λέμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο ειδικοί όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της ενέργειας και αυτό να εγκριθεί σε επίπεδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι τώρα στην πυρηνική ενέργεια. Όσον αφορά λοιπόν την πυρηνική ενέργεια, η Προεδρία θα ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε μια οδηγία Europe Atom όπου θα προβλέπονται οι προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων από την ακτινοβολία. Εδώ πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα από τα διάφορα τεστ αντοχής, stress test που έχουμε κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά την ασφάλεια. Και αυτό όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις χώρες που γυρνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να έχουμε ιδιαίτερα ψηλέ προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο μέσα σε αυτήν. Για τα θέματα ενέργειας θα τελειώσω με το εξή. Θέλουμε να αλλάξουμε τη ρητορική που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στις οικονομίες με χαμηλό αποτύπωμα ε, διοξιδίου του άνθρακα, αλλά πρέπει να δούμε και την οικονομική πτυχή. Με λύσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στο να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίε που έχουμε μπροστά μας. Γιατί αν μιλάμε μόνο για το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, μιλάμε μόνο για το άνθρακα. Ενώ αν μιλάμε γενικότερα για χαμηλέ εκπομπές, δεν μιλάμε μόνο για τον άνθρακα, μιλάμε και για τις άλλες ε, μορφές καυσίμων που χρησιμοποιούμε. Πάντα με ασφάλεια εφοδιασμού βέβαια. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καλύτερη χρήση της ενέργειας. Για παράδειγμα, αν ε, μιλάμε για την χρήση για τη χρήση χιστόλιθου πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί χρησιμοποιώντας δύο φορές παραπάνω. Πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις αντλίες θερμότητας έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αντιγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το δικό μας μότο λοιπόν είναι χαμηλές ε, εκπομπές, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Γι' αυτό θα συνεργαστούμε και με τη βιομηχανία και με διεθνείς οργανώσεις. Έχουμε ακούσει και τη, τα, περί της τελευταίας έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας που αναφέρεται σε αλλαγές και στην οικονομία. Η έκθεση αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας ε, δείχνει και πώς να τροποποιήσουμε την οικονομία μας έτσι ώστε να καταλήξει σε χαμηλές εκπομπές διατηρώντας όμως την ανταγωνιστικότητά της. Όσον αφορά τώρα τη βιομηχανική πολιτική, εδώ θέλουμε να γίνει μια συζήτηση στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ευέλικτε πρωτοβουλίες. Πώς θα δούμε δηλαδή τη βιομηχανική πολιτική στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, πώς θα δούμε την καινοτομία, πώς θα δούμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων και των πηγών. Γι' αυτό και υπάρχει ένας οδικός χάρτης για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο μιας άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα, δηλαδή. Το Συμβούλιο αυτό θα γίνει στο Σόμποτ στις 21 και 22 Ιουλίου. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω επίσης ότι στόχος μας είναι η βιομηχανική πολιτική να επικεντρώνεται στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη όμως κάθε φορά τις επιπτώσεις που έχει η πολιτική μας στην ανταγωνιστικότητά μας. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα από την κρίση και να αντιληφθούμε την μη και πραγματική αλήθεια που είναι ότι όταν έχουμε παραγωγή ή απασχόληση μπορούμε να έχουμε και οικονομική ανάπτυξη. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Περί αυτού πρόκειται και περί του να προστατεύσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Τώρα έρχομαι σε άλλε δραστηριότητες οι οποίες θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Το Συμβούλιο 29 και 30 Σεπτεμβρίου θα έχουμε Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα. και στη συζήτηση εκεί θα προσπαθήσουμε να εγκρίνουμε και κάποια συμπεράσματα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τέλος, θέλω να σας πω πως οι πρωτοβουλίες αυτές θα ολοκληρωθούν με συζήτηση. Θα συζητήσουμε για εμβληματικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια. Περιμένουμε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια. Πάντως η προετοιμασία για τα συμπεράσματα θα ξεκινήσει με την ομάδα εργασίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα τον Οκτώβριο ή και αρχές Νοεμβρίου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την Προεδρία μας με ενθουσιασμό. Όπως ξέρετε, τον Οκτώβριο έχουμε κοινοβουλευτικέ εκλογές στην Πολωνία. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάπως λεπτά τα πράγματα για την Προεδρία μας. Δεν λέω ότι είναι mission impossible, ε, ότι είναι αδύνατο να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας, απλώς είναι λίγο λεπτό το θέμα. Όπω είπε και ο Πρωθυπουργό μα, μπορούμε να ξεχάσουμε τι διακοπέ φέτο το καλοκαίρι εμεί. Χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ. Πάντω, όπως και να έχουν τα πράγματα, το Σεπτέμβριο θα συνεχίσουμε με τη δουλειά μας και ελπίζουμε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας αποφασιστικής σημασίας μήνας για πολλά από τα θέματα που μας απασχολούν. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βασίζομαι στη δικιά σας στήριξη και στη δικιά σας συνεργασία. Θέλουμε την εμπειρία σας, μας είναι πολύτιμη. Εσείς δουλεύετε σε αυτό το τομέα εδώ και καιρό, συνεχώς και σίγουρα μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ξέρετε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχετε τις δικές σας ευαισθησίες, τις δικές σας εμπειρίες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε την βοήθεια και τη συνεργασία σας και ελπίζουμε η Προεδρία μας να προσφέρει νέα όθηση υπέρ της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και όταν είναι κανείς επιμελής, αυτό συνήθως αποδίδει αποτελέσματα. Τώρα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στους ομιλητές αν περιορίσουν τις ερωτήσεις τους σε ένα το πολύ δύο λεπτά για να υπάρχει χρόνος να απαντήσει ο κύριος Παύλαξ στο τέλος. Ξεκινάμε με τον κύριο Βέμπα. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω κιόλας και για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας Πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε την ενεργειακή, ενεργειακή πολιτική και την ασφάλεια προμήθειας. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι το πιο σημαντικό. Ήθελα όμως να κάνω μια παρατήρηση για την πρόταση που έγινε από πλευράς της Επιτροπής ε, να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα ε, GMES εκτός του επόμενου χρηματοδοτικού πλαισίου της κοινότητας 2014-2020. Αυτό παραβιάζει τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στο πρόγραμμα αυτό, το GMS, να σταματήσει λόγω ακριβώς του ότι δεν θα υπάρχει εγγυημένη χρηματοδότηση και κινδυνεύουμε απλώς να ε, κατασπαταλήσουμε τις ε, ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει και που ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία εκ των οποίων το 1 τρίτο δόθη από το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και τα υπόλοιπα από τον Οργανισμό το, ε, Διαστημικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα να ρωτήσω τι κάνετε για αυτό το, τόσο μεγάλο πρόγραμμα για την, ε, το διαστημικό έτσι ώστε να μην ε, το εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα αυτό και να παραμείνει εν ζωή. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις ε, κύριε Υπουργέ. Η πρώτη ερώτηση αφορά την εφαρμογή της έκθεσης από μερικού μήνες για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική. Ένας Γερμανός συνάδελφος, ο κ. Μπερνλάνγκε ήταν ο εισηγητής. Ήθελα να ρωτήσω τι προτίθεστε να κάνετε για να βοηθήσετε να, διο... να παραμείνουν οι θέσεις απασχόλησης στην παραδοσιακή βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εκεί χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερον, μιλήσατε για ενεργειακή πολιτική, μιλήσατε για εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, με την ανάγκη να παράγουμε όμως περισσότερη ενέργεια. Θα χρησιμοποιήσουμε ούτως ή άλλως ε, περισσότερες, ε, το περισσότερο άνθρακα για την ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όμως με την πολιτική και την τεχνολογία συγκράτησης και του διοξιδίου του άνθρακα και αποθήκευσής του μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Επομένως θα έπρεπε η Πολωνία να πιέσει περισσότερο έτσι ώστε να υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόγραμμα ε, συγκέντρωσης και αποθήκευσης ε, του διοξιδίου του άνθρακα, έτσι ώστε να μπορεί να ε, παραμείνει εν ενεργεία ο τομέας αυτός. Ευχαριστώ, κυρία Έκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο. Εδώ είμαι, στο μέσο μου. Ευχαριστώ. για τον οδικό χάρτη για την ανάργεια. Με ανησυχεί ιδιαίτερα γεγονός, το γεγονός ότι μετά το τελευταίο Συμβούλιο Ενέργειας η απόφαση του Επιτρόπου να ε, το Δεκέμβριο με την Νότια Αφρική Τη Επιτρόπου μάλλον, ε, μας αναγκάζει να υιοθετήσουμε μια πλατφόρμα, διότι αλλιώ πώς θα προχωρήσουμε. Ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας της προμήθειας ε, της ενέργειας. Χρειαζόμαστε κάποιες αποφάσεις, όπως είπατε και εσεί, είναι θέμα προτεραιότητα. για να υπάρχουν καλέ συνθήκε εργασία, αν θέλετε. Δεύτερον, για την αποτελεσματικότητα των πόρων ενέργειας. Πώς το βλέπετε να διαμορφώνεται το θέμα. Και τρίτον, μία συμβουλή. Ελπίζω ότι στον τρίλογο θα λειτουργήσει τόπος η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή με ανοιχτή εντολή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και τους φακέλους τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω, λέει η κυρία Ριβάζη, τον Υπουργό. Ε, είμαστε στην Πολωνία με την αντιπροσωπεία μας και ε, εκεί μιλήσατε για μία ενεργειακή στρατηγική ε, που θα έχει λιγότερο άνθρακα, θα χρησιμοποιεί λιγότερο άνθρακα. Αυτό, πολύ καλό αυτό όμως. Ταυτόχρονα όμως έχετε πολύ άνθρακα και θέλετε να αναπτύξετε, να αναπτύξετε ε, μια πολιτική, μια βιομηχανία παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιώντας ε, σχιστόλιθο. Όμως ο σχιστόλιθος παράγει πολύ μόλυνση, μεγάλη μόλυνση. Και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η εγγύηση την οποία προσφέρετε στους πολίτες που, τον οποίο θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ε, σε σχέση και με, τις, ε, με τον μεγάλο αριθμό αδειών που έχετε δώσει και υπάρχουν ε, εξορίξεις που, γίνεται, που γίνονται, πολλές εξορίξεις γίνονται αυτή τη στιγμή, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. Ποιος θα πληρώσει, ποιος θα καθαρίσει την, τον υδροφόρο ορίζοντα. ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε στο Κοινοβούλιο κύριε Παύλα και με μεγάλη χαρά σας ατενίζω. Όλα αυτά τα οποία είπατε έχουν μεγάλη σημασία και στην Επιτροπή μας θα βρείτε πραγματικούς συμμάχους για να σας υποστηρίξουν στις δραστηριότητες που θέλετε να αναλάβετε. Σήμερα μόλις ψηφίσαμε μια έκθεση για, την, ε, για τον κανονισμό REMIT και αυτό ανοίγει το δρόμο έγκρισης σε πρώτη ανάγνωση. Χθε ακούσαμε ότι η κυβέρνησή σας θέλει να ασχοληθεί για τον κανονισμό benchmark βαθμονόμησης για το φυσικό αέριο. Αυτό είναι μια πολύ καλή απόφαση. Είναι πολλοί οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρούν ότι είναι σωστή η μέρημνά σας για τα ζητήματα αυτά και πιστεύουμε ότι το να βασίσουμε την αγορά διοξιδίου του άνθρακος χαμηλού μάλλον, χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος μόνο στο φυσικό αέριο είναι κάτι το οποίο είναι άδικο για πολλές χώρες. Μπορείτε όμως να μας πείτε περισσότερο για την πρωτοβουλία αυτή της Πολωνίας, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του εγχειρήματος σε σχέση με την απόφαση που έχετε λάβει. Κύριο Μπρεζίνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον κύριο Υπουργό και στην Πολωνική Προεδρία σε σχέση με την ε, πυρηνική έρευνα για την πυρηνική ενέργεια. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ένα πρόγραμμα για έρευνα στον πυρηνικό τομέα. Αλλά τίθεται το θέμα του αν θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτού του προγράμματος και της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, της σύνδεσης με τα δίκτυα. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η Πολωνική Προεδρία θέλει να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια και την ενέργεια σύνδεξης, όπως στην περίπτωση του προγράμματος JET στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν θα μπορέσουν να περατωθούν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια ακόμα της Πολωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίρεκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και έχω να κάνω ορισμένα ερωτήματα, αλλά θα, είμαι... θα αυτοπεριοριστώ σε ένα ερώτημα και μονάχα ως μηχανικός, εσείς προσπαθείτε να είσαστε ορθολογικός ε, για τα θέματα της ε, αποδοτικής χρήσης ενέργειας και αναφερθήκατε και σε εκπομπές αριών του θερμοκήπιου. Πώς βλέπετε τις δυνατότητες να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ δεν συμφωνώ με ένα προλαλήσαντα. Νομίζω ότι η συγκράτηση και αποθήκευση του άνθρακα είναι ένα σημαντικό θέμα. Πώς το βλέπετε αυτό, θεωρείτε ότι θα μπορέσει αυτό να ληφθεί υπόψη επαρκώς στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Καρβάλιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας και για όλες αυτές τις εκτενείς εξελίξεις, εξηγήσεις που μας δώσατε. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όλο το πρόγραμμα αυτό συγκέντρωσης, αποθήκευσης ε, του άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούμε να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει διότι η χρήση του άνθρακα ούτως ή άλλως αυξάνεται και υπάρχει ούτως ή άλλως η τεχνολογία σε πιλωτικό επίπεδο και η Ευρώπη έχει χρηματοδοτήσει ε, πολλές αρκετές ε, αρκετά project σε ε, πραγματική κλίμακα. Ένα, μια εγκατάσταση βρίσκεται ούτως ή άλλως στην Πολωνία, όμως παρουσιάζονται κάποιες τεχνολογίες, ε, κάποιες δυσκολίες, όχι τεχνολογικού χαρακτήρα, αλλά συγχρηματοδότησης. Επομένως, εσείς σαν Προεδρία, ε, τι προτίθεσα να κάνετε, έτσι ώστε αυτά τα project να προωθηθούν, για να που θα αποδείξουν και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας. Επίσης, όσον αφορά την ε, προσαρμογή των, ε, την ενεργειακή προσαρμογή των υπαρχόντων κτηρίων, γιατί ώστε να γίνουν από πιο αποτελεσματικά από ενεργικής πλευράς. Υπάρχει ένα ταμείο ήδη, αλλά λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα του όλου θέματος ε, δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε πλήρως. Επομένως, εσείς τι πρέπει να κάνετε όσον αφορά αυτή τη ε, διαμόρφωση των κτηρίων για να γίνουν πιο αποτελεσματικά ενεργειακά. Ε, κυρία Ήμπνερ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε <clears throat> και εγώ θέλω να χαιρετήσω τον ε, κύριο Παύλα και εδώ χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας. Από αυτά τα οποία γνωρίζουμε, από αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα, έχετε φιλόδοξα σχέδια, αναφερθήκατε σε ένα νέο κανονισμό για την ε, ενεργειακή απόδοση, για τον κανονισμό Ρέμιτ επίσης αναφερθήκατε και επίσης για μια νέα οδηγία που αφορά υψηλά επίπεδα ασφαλείας στην χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Όλα αυτά είναι πολύ φιλόδοξοι στόχοι. Στην Ευρώπη όμως έχουμε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα και κάποιες αποκλήσεις απόψεων για το σωστό ενεργειακό μείγμα και για την αναδιάρθρωση αυτού του μείγματος ώστε να είναι προς όφελος όλων. Ποια είναι η δική σας πρόταση από την πλευρά της Πολωνίας. Θα βασιστείτε στην πυρηνική ενέργεια, θα εξακολουθείτε να ε, υποστηρίζετε την συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Πολωνίας και εξετάζετε στο Συμβούλιο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει αρρωγή προς τα κράτη-μέλη. Γιατί πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας και γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες θα έχουν δυσκολία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Δεν έχουν επιτύχει τους στόχους που <clears throat> είχαν θέσει στον εαυτό τους για τις εναλλακτικές ενέργειες. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν σε επίπεδο κρατών μελών και ευρωπαϊκό το θέμα του ενεργειακού μείγματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του. Κατανοώ βέβαια ότι είναι πάρα πολύ πλούσια η μέση διάταξη της Πολωνικής Προεδρίας και πολύ φιλόδοξη. Νομίζω ότι η υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα πρέπει να αποσκοπεί στο να υπάρχει καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, στον ενεργειακό χώρο. Εγώ θα ήθελα να έχω και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε σχέση με την ε, αντιμετώπιση που υπάρχει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οικονομικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τι θα πράξετε σχετικά. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των ευρεσιτεχνιών και εκεί έχουμε θέματα, θέματα τα οποία είναι ε, εκρεμή. Νομίζω ότι είναι σημαντικές ευρεσιτεχνίες για την καινοτομία. Ένα τρίτο θέμα σε σχέση με την τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πρότυπα θα πρέπει να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα τελευταία φράγματα τα οποία μένουν στο επίπεδο της ε, εσωτερικής αγοράς για την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, προϊόντων και εμπορευμάτων. Και ένα τελευταίο ακόμα ερώτημα. Στην ε, παρουσίασή σας αναφερθήκατε στην ενεργειακή πολιτική λέγοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και διμερείς λύσεις για τα ενεργειακά προβλήματα. Τι ακριβώς εννοούσατε. Νομίζω ότι η δική μας στρατηγική βασίζεται περισσότερο στο να υπάρχει ένας ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην παρεμβαίνουν πολιτικές ε, θεωρήσεις και στοιχεία. Ο κ. Γκρίτσος είναι ο τελευταίος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι έχετε δυσκολίες με το όνομά μου, αλλά τα πράγματα βελτιώνονται σιγά σιγά. Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία σας και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Και επίσης να σας ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει για την Επιτροπή μας. Θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Έχουμε ένα θέμα να αντιμετωπίσουμε με την απόσυση από την πυρηνική ενέργεια του γείτονά μας, της Γερμανίας, η οποία μέχρι το έτος 2022 θα κλείσει όλους τους πυρηνικούς σταθμούς. Ενώ γνωρίζουμε ότι Περίπου το 1 τέταρτο της παραγόμενης ενέργειας στη Γερμανία προέρχεται από πυρηνικούς σταθμούς. Θέτω λοιπόν το ερώτημα τι θα σημάνει αυτό γενικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Ποια είναι η δική σας θέση σχετικά σε σχέση με τη χρήση ενός νέου ενεργειακού μείγματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι για τη χρησιμοποίηση των, των εναλλακτικών συγγνώμη ενεργειών. Εντάξει, ναι αλλά αυτό είναι ένα ανεξερεύνητο τοπίο ακόμα. Είναι ανάγκη να δούμε λοιπόν με ένα διαφορετικό τρόπο όλους αυτούς τους νέους φορείς εναλλακτικής ενέργειας. Επίσης αναφερθήκατε και στην τεχνολογία καθαρής καύσης άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα νέο μάτι στην Ευρώπη. Επίσης, τα θέματα των αγωγών φυσικού αερίου και της διασύνδεσής της, τα προβλήματα ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντος που ανέφερε η κυρία Ριβάζη. Υπάρχει επίσης και η δημιουργία νέων υποδομών που μπορούν να ε, χρησιμοποιούν το μεθάνιο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέροντα που λέτε. Σα ευχαριστώ πολύ και δίνω τώρα πάλι το λόγο στον κύριο Παύλα. E, e, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πολλές και διάφορες οι ερωτήσεις σας. Και θα ήθελα να κάνω καταρχάς ένα γενικό σχόλιο, το οποίο σχετίζεται με την ενεργειακή αλλά και με την βιομηχανική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφώσουμε το γενικότερο πλαίσιο σωστά. Εάν τεθούν δηλαδή οι αρχές με σωστό τρόπο, τότε οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Επίσης θα πρέπει να ε, έχουμε κατά νου και την αρχή της επικουρικότητας, διότι και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και κάτι άλλο. Σε πάρα πολλούς τομείς ε, που σχετίζονται με τεχνικές πτυχές, προδιαγραφές κτλ, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα εάν είχαμε υιοθετήσει κανονισμούς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα εφαρμόζαμε τις ίδιες προδιαγραφές. Για άλλα θέματα όμως που άπτονται πολιτιστικών πτυχών πρέπει να υιοθετήσουμε άλλες λύσεις. Όμω, θα πρέπει τα βασικά να ρυθμίζονται με κανονισμούς έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα ίδια παντού. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο πακέτο ε, το ενεργειακό. Υπάρχει δυνατότητα μεταβατικών περιόδων. Υπάρχει, είναι το περίφημο 10 γάμα, το άρθρο από το περίφημο 10 γάμα και στα, συμβούλια, στα συμπεράσματα συγγνώμη, του Συμβουλίου υπάρχει μία ρήτρα που λέει ότι οι εξαιρεσει αφορούν τις εγκαταστάσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό υιοθετήθηκε το 2008. Το 2011 τώρα, στις ε, οδηγίες που δίνει, κατευθύνσεις οδηγίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει μια παρόμοια διάταξη που αναφέρει ε, τα εξή ότι πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό πώς να το ερμηνεύσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά τα όσα είχαμε αποφασίσει το 2008. Ποιες είναι οι συνέπειες τώρα όλων αυτών. Είναι ότι οι επιχειρηματίες δεν προχωρούν σε επενδύσεις, δεν υπάρχει νομική σαφήνεια όσον αφορά τον κανονισμό αυτό. Και Αυτά πρέπει να έχουμε κατά νου για να επιστήσουμε την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων σε κάποια σημαντικά θέματα. Δηλαδή, αν αλλάξουμε την αποτελεσματικότητα των εγκαταστάσεων, δηλαδή ε, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ε, ενέργειας ε, και από 33% πάμε στο 50%, τότε οι εκπομπές θα μειωθούν κατά, κατά το 1 τρίτο. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει νομική σαφήνεια. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους project δηλαδή, θα πρέπει όλες οι λεπτομέρειες να είναι ε, ξεκαθαρισμένες. Ο κύριος Βέμπερ τώρα μίλησε για, το, για την αεροδιαστημική ε, και την πολιτική μας για το διάστημα. Ε, ένας από τους στόχους της Πολωνικής Προεδρίας, και αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από την δημοσίευση του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, είναι να συζητηθεί το θέμα αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών και αφού εντοπίσουμε τα πιο σημαντικά ε, θέματα, τα οποία προφανώς θα συνεχίσουν να, να συζητώνται και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Δανίας. Προφανώς όλα αυτά τα, όλες αυτές οι επενδύσεις που έχουν γίνει στα κοινά διαστημικά προγράμματα δεν θα πρέπει να ε, χαθούν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει κάποια εφαρμοστικά μέτρα γιατί οι επενδύσεις αυτές και τα project αυτά μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο στο διάστημα αλλά και σε πιο καθημερινά θέματα που αφορούν άμεσα τον πολίτη. Επίσης ήθελα να τονίσω, να υπενθυμίσω ότι θα υπάρξει μια συνάντηση των διευθυντών για την ενέργεια στην Πολωνία όπου θα συζητηθεί ο αντίκτυπος της γερμανικής απόφασης για το πάγωμα των πυρηνικών εργοστασίων στην Γερμανία. Επίσης θα συζητήσουν και τα θέματα ε, των πηγών ενέργειας ε, που, ε, που έχουν λιγότερες εκπομπές. Αυτή η συνάντηση γίνει στον Μπελχάτοφ. Γιατί τώρα θα γίνει αυτό, διότι εκεί υπάρχει ένα, μια μονάδα συγκράτηση και αποθήκευσης άνθρακα εκεί, από τις πιο σημαντικές μονάδες που έχουμε. Και αυτό γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα. Βέβαια, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι παρά τον μεγάλο ενθουσιασμό, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν πολλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς δεν θα το είχαμε υλοποιήσει αυτό το project αν δεν υπήρχε η κοινοτική συγχρηματοδότηση. Δεν θα ήταν βιώσιμο ένα τέτοιο project. Γι' αυτό θα πρέπει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο, να ε, κοστολογήσουμε συγκεκριμένα το κόστος παραγωγής ε, αυτών των μονάδων εγκατάστασης, αυτών των ε, μονάδων συγκράτησης και αποθήκευσης άνθρακα. και το πρόβλημα είναι ότι συναντάμε πολλές φορές και την ε, αντίδραση των πολιτών, αυτών που κατοικούν στις περιοχές αυτές, διότι ε, τους λέμε ότι θα αποθηκεύεται το διοξείδιο άνθρακα, δεν είναι σίγουροι. Γι' αυτό θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις, ε, την ενέργεια. Υπάρχουν και θέματα μεταφορών τώρα, μεταφορών ας πούμε, που άπτονται, μεταφορές που άπτονται του, του, της ηλεκτρικής ενέργειας, ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί για το 10%. Δηλαδή 10% χρησιμοποιείται για τις ε, μεταφορές, ενώ 40% της ενέργειας χρησιμοποιείται για την μεταφορά του αυτοκινήτου. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αποθήκευση της ενέργειας. Η ενέργεια αυτή δηλαδή αποθηκεύεται όταν δεν χρησιμοποιείται και η ενέργεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι στο δίκτυο. Κάποιοι Ιάπωνες ερευνητές λένε ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί 3% μόνο για τη μετακίνησή του και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιείται για την μετακίνησή του. Αποθηκεύεται. Όταν ερχόμαστε στα κτίρια τώρα και την απόδοση των κτιρίων και εκεί έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη με την μόνωση των σπιτιών, με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σπίτια, δημιουργούνται και θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα άλλο θέμα αφορά τον οδικό χάρτη για το 2015 και τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος για την ε, αύξηση ε, του στόχου από 20-25%. Εδώ η Πολωνία, η στόχη για το 2050, ε, η Πολωνία πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν ειλικρινείς συζητήσεις ε, για τις λύσεις αυτές. Θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη μας ε, και τους στόχους μείωσης. Θα πρέπει να γίνουν δηλαδή ε, συνολικές συζητήσεις και να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να επιβληθούν τέτοιου είδους αυστηρές διατάξεις στην βιομηχανία εάν δεν έχουμε και ορατά αποτελέσματα πλεονεκτήματα για την βιομηχανία. Ένας επιφανής οικονομολόγος, ο οποίος επισκέφθηκε την Πολωνία και μίλησε για την ε, ενέργεια και την ενεργειακή πολιτική, ε, είπε ότι η, από το 20 για να πάμε στο 25% αυτή η διαφορά είναι οι εκπομπές της Κίνας για μία εβδομάδα και μόνον. Άρα χρειάζεται πολλή ε, συζήτηση και, να, και χρειάζεται και συμφωνία, γενική συμφωνία, εάν ε, πρέπει να δράσουμε. Απ' την άλλη πλευρά, η, Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να υιοθετηθεί αυτή η, η αύξηση του στόχου από 20-25%. Στην Πολωνία θα γίνει μια συνάντηση των 20 ε, μεγάλων παραγωγών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης ε, καλέσαμε εκπροσώπους της τσιμεντοβιομηχανίας και παραγωγής αλουμίνας και συζητήσαμε την ανάγκη να ορίσουμε συγκεκριμένα όρια ανατομής έτσι ώστε να μην υπάρχει ένας ανταγωνισμός ε, ο οποίος θα οδηγούσε στην χρήση βρώμικης τεχνολογίας. Και ούτως ή άλλως είναι πολύ απτά τα αποτελέσματα ε, εάν αυτές οι βιομηχανίες ε, αλουμίνας, τσιμεντοβιομηχανίες, τα χαλιβουργία μειώσει τις, τις εκπομπές, μειώσουν τις εκπομπές τους και νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σφαιρική απόφαση. Δεν θα πρέπει μονομερός να προχωρούμε. Επίσης, όσον αφορά τα guns, τα gas benchmarks, ε, ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία στο παρελθόν οι σοβιετικοί μηχανικοί είχαν παράγει, είχαν φεύρει μία λεπίδα ξυριστική. Κάποιος έβαζε το κεφάλι του σε μία τρύπα και μετά έβγαινε και ήταν ξυρισμένος. Του είπαν όμως κάποιοι ότι ναι, αλλά ξέρετε, διαφορετικό πρόσωπο, διαφορετικό κεφάλι έχει ο καθένας, τι θα γίνει. Α, δεν πειράζει, το πρόβλημα θα παρουσιαστεί μόνο την πρώτη φορά. Μετά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε εδώ, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ χώρε, διαφορετικέ ανάγκε, διαφορετικέ ιδιαιτερότητε. Λοιπόν, εμεί δεν είμαστε σε θέση να το διακινδυνεύσουμε έτσι όπω ε, η σοβιετική μηχανική. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του άνθρακα και τα να σας πω ότι... Shell. Λοιπόν, τώρα γι' αυτό το, το, το αέριο από τους σχιστόλιθους, τι να σας πω, εσείς ε, χαίρομαι που είδατε ότι υπάρχει και κάτι που είναι πιο επικίνδυνο από τον άνθρακα. Ε, πάντως, ε, προφανώς θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη μας και την ε, ενεργειακή προμήθεια, αλλά και, την, και, το, και, το, και το περιβάλλον. εάν είχαμε μία τεχνολογία αποτελεσματική όσον αφορά την συγκράτηση και την αποθήκευση του άνθρακα, προφανώς ο άνθρακας θα ήταν τόσο περιβαλλοντικά φιλικός όπως και άλλες πηγές ε, ενέργειας. Τώρα, για το, φυσικό, για το, το αέριο που παράγεται από το σχιστόλιθο, προφανώς ε, κάθε πηγή ενέργειας, αν θέλετε, χρειάζεται και την ε, δική της τεχνολογία έστω και αν βρούμε αέριο από το σχιστόλιθο, θα πρέπει, ε, δεν είναι σίγουρο μάλλον ότι μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Εάν δεν είναι ασφαλής η χρησιμοποίηση και αν δεν υπάρχει κίνδυνος ε, μόλυνσης ε, του υδροφόρου ορίζοντα από το μεθάνιο, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Εδώ υπάρχει ένας άλλος παρόμοιος κίνδυνος για τον άνθρακα διότι η εξόριξη του άνθρακα και η χρησιμοποίηση του άνθρακα δεν είναι μόνο ε, προβληματική για το περιβάλλον, μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα, προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά. Ο κύριος Σιμάνσκι αναφέρθηκε στην οδηγία Ρέμετ και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η οδηγία αυτή εισάγει λύσεις ε, που μπορεί να είναι αποτελεσματικές ε, όσον αφορά την αγορά. Γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου πολλές φορές ε, καθυστερούν. Όμως η διαφάνεια επιτρέπει οι εμπλεκόμενοι να, έχουν τις ίδια, να γνωρίζουν τι συμβαίνει, να έχουν μια κοινή άποψη αν θέλετε. Κάποια στιγμή όταν είχα μιλήσει για την διαφάνεια με κατηγόρησαν ε, ότι είμαι αντίθετος ε, στην ε, κοινή αγορά. Εγώ είπα όχι, ίσα ίσα. Για να υπάρχει κοινή αγορά πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια. Πρέπει να έχουμε όλοι τις ίδιες πληροφορίες. Και αυτή η οδηγία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πολύ σημαντική για την ενεργική πολιτική. Τώρα όσον αφορά την πυρηνική έρευνα. Η Κομισιό θέλει να αλλάξει πέντε οδηγίες ε, για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας, ε, για την πυρηνική ενέργεια και την πυρηνική έρευνα. Και η Κομισιόν θέλει να συγκεντρώσει αυτές τις πέντε οδηγίες σε μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μία σωστή ισορροπία. Όταν έχουμε πέντε προτάσεις ε, νομοθετικού περιεχομένου, έχουμε προφανώς μία δυσκολία. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν έχουμε μία και μόνη νομοθετική πρόταση, πρέπει να είναι σωστή, να είναι πολύ καλή πρόταση. Και ελπίζω ότι οι οδηγίες αυτές, η οδηγία αυτή μάλλον θα υιοθετηθεί ε, άμεσα, διότι πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος απαιτεί άμεσες ε, απαντήσεις, χρειάζονται και δοκιμασίες αντοχής, Θέλω να τονίσω ότι θέλουμε όλες αυτές οι λύσεις που αφορούν την ασφάλεια να εφαρμοστούν. Δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι λύσεις και τα μαθήματα, τα διδάγματα που αποκομίζουμε από τα τεστ αντοχής, τα stress test, θα πρέπει να επεκταθούν και στους ε, γείτονές μας. Κύριε Γκέρακ, αναφερθήκατε στην τροποποίηση του ενεργειακού μείγματος ή του κλιματικού πακέτου μέτρων, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι λύσεις αυτές να έχουν κάποια σταθερότητα στο χρόνο. Είναι κεφαλαιόδες το θέμα αυτό. Θα πρέπει βέβαια να ενημερώνουμε και να επικαιροποιούμε αυτές τις λύσεις συχνά. Δεν μπορεί μία ιδέα να επικρατεί πάντα πάνω στην κοινή λογική αν αποδειχθεί ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι πολυδάπανες, όπως παραδείγματος χάρη συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακα και για τη δική μας την ε, εγκατάσταση στο Μπελχατούπ οι μελέτες λένε ότι χρειάζονται, θα κοστίζει περίπου 60 ευρώ για να αποθηκεύσουμε ένα τόνο άνθρακα. Ενώ μία μεγαβατόρα, ένα μεγαβάτ ώρα, είναι περίπου 60 ευρώ επίσης. 50 ευρώ στην πραγματικότητα στη δική μας περιοχή. Βλέπετε λοιπόν ότι κοστίζει περίπου 1 προς 1 η παραγωγή ενέργειας με την χρησιμοποίηση της συγκράτησης και αποθήκευσης άνθρακα. Αυτό θα παίξει και κάποιο μεγάλο ρόλο για το κόστος της λειτουργίας αυτής της εγκατάστασης και αυτό θα αύξανε κάθετα τις τιμές της ενέργειας. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν για λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες από οικονομική άποψη. Και πάρα πολύ σύντομα για το ενεργειακό μείγμα θα ήθελα να πω το εξής. Η θέση μας για, την, ε, για τα κριτήρια, για τα benchmarks είναι η εξής. Η Πολωνία έχει εστιάσει την θέση της στο ότι το ενεργειακό μείγμα βάσει και των συνδικών καθορίζεται σε επίπεδο κρατών μελών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να τύχουν σεβασμού αυτές οι βασικές αρχές. Γιατί έχουμε κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την ε, εξόριξη, την υπεράκτια εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου όπου και σε αυτή την περίπτωση εμπλέκεται αποκλειστικά η αρμοδιότητα και η ευθύνη των κρατών μελών. Η θέση λοιπόν της Πολωνίας για όλα αυτά είναι η εξή λέμε ότι θα πρέπει να <clears throat> προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών. Έχουμε και κάποιους στόχους για την πυρηνική ενέργεια, αλλά μετά από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Γερμανία θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα, να υπάρξει μια διαδικασία αναθεώρησης και να δούμε αν έχει πιο πολύ νόημα να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να συγκρίνουμε διαφορετικά σενάρια, διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις. Γενικά όμως τα σχέδια της Πολωνίας δίνουν έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια ως, οι πιο, ως τους πιο σημαντικούς παράγοντες αλλαγής του ενεργειακού μείγματος. Και βέβαια, δεν, για τις ευρεσιτεχνίες δεν έχουμε πετύχει πολλά πράγματα μέχρι στιγμής, αλλά μετά από 30 χρόνια επιτέλους είναι καιρός να λειτουργήσει και η ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία. Κατανοούμε τα επιχειρήματα των Ιταλών και των Ισπανών, τους ακούμε προσεκτικά τα επιχειρήματα που αναπτύσσουν. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει και δική του συμφωνία και προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ευρωστεχνία. Για τα πρότυπα επίσης θεωρώ ότι τα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόζονται με τυποποιημένης μορφής κανονισμούς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να αντλήσουμε ταχαίως ωφέλη από την ενική αγορά. Και εδώ μια συμβολική εμπειρία μπορεί να είναι η ενοποίηση των ε, βυσμάτων για τα κινητά τηλέφωνα. Να είναι δυνατόν να έχουμε όλοι <coughs> το ίδιο είδος φορτιστού για τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι κάτι πολύ απτό και κάτι που κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών μας και αυτό θα μπορούσε να προκύψει και από, θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση του κόστους των ε, κινητών τηλεφώνων, γιατί ο καθένας πάντα πρέπει να ψάχνει να βρίσκει τον κατάλληλο φορτιστή για το τηλέφωνό του. Ένα ακόμα θέμα το οποίο δεν ανέφερα. Ο κύριος Γκριπς έθεσε ένα ερώτημα το οποίο το απήντησα εν μέρος που είναι οι συνέπειες της γερμανικής απόφασης για την ε, απόσυρση από την χρήση πυρηνικής ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν Εν κατακλείδη να σας πω ότι η Προεδρία είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας, με τους εισηγητές σας και βασιζόμαστε και στις προσωπικές επαφές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κατεπήγον, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θέλω να σας ζητήσω να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες των Πολωνών συναδέλφων που είναι μέλη της Επιτροπής σας. Εμείς έχουμε λοιπόν απόψεις στην Πολωνία που είναι εδρεωμένες, ακόμα και η αντιπολίτευση έχει απόψεις που σε μεγάλο βαθμό είναι κοντά στις δικές μας. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις υπηρεσίες των Πολωνών Ευρωβουλευτών, θα μπορέσουν να μεταλαμβαδεύσουν τις απόψεις σας. Βασιζόμαστε λοιπόν και στη δική σας εμπειρία και για να το πω αυτό με πιο συμβολικό εμβληματικό τρόπο προχωρούμε προς μια διαδικασία πράσινης ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας, μια βιώσιμη ανάπτυξη και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να συνυπολογιστούν όλοι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συγχρόνως με τους οικονομικούς παράγοντες. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ό,τι περνάει από τη δική μας πλευρά, ώστε να είμαστε από την πράσινη μεριά του δάσους και όχι από την άλλη. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε καταφέρει να απαντήσετε πάρα πολλά και διαφορετικά ερωτήματα. Αυτό είναι όμως και το στοιχείο των συζητήσεων, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, τα απαντήσατε με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Πραγματικά θα μας δώσει μεγάλη ευχαριστήση να συνεργαστούμε μαζί σας για όλα αυτά τα πολλαπλά